Πρόεδρος, συνάδελφε, συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. Αρχίζουμε. Καλώς ορίσατε. Στη συνέχεια των θερμοδιακοπών. Πρώτα-πρώτα να εγκρίνουμε την μέση διάταξη. Αν κανείς δεν έχει κάποια ένσταση, τότε ευθύ αμέσω να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 4. Το 4 είναι. Όχι, το 6. Το 6 διορθώνει η πρόεδρο. Το 6 διάταξη είναι η μεταρρύθμιση του συστήματο ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπρέσο έχει ένα πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα μα σήμερα, γι' αυτό να τη δώσουμε το λόγο ευθύ αμέσω και τα άλλα να τα συζητήσουμε μετά. Κύριε Μπρέσο, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και στα Ιταλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια γνωμοδότηση όχι, δεν είναι ε, έκθεση βέβαια, είναι αυτή. Στη συνέχεια της έκθεσης Λεβαντόφσκι και Ντεπρέ όσον αφορά τους ιδίους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησε τις προτάσεις ε, οι οποίες υπευλήθησαν ε, από την ομάδα ψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίσης και σχετικά έγγραφα εργασίας αυτά, τα οποία έχουν σχέση με το έγγραφο. Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση ε, αφορά την Επιτροπή των Προϋπολογισμών, κυρίως αρμοδία, και περιορίζεται στο να ε, θυγεί τα ζητήματα θεσμικής, συνταγματικής φύσεως. Αυτά τα οποία από των δικών μας του ενός Επιτροπής και επίσης υπενθυμίζεται ότι έχουμε δύο άρθρα της Ένωσης που ορίζουν πώς θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 310 πρώτα πρώτα που δεν μπορεί να έχει κάποιες πράξεις η Ένωση να τις εκδίδει που να έχουν σημαντικές πτώσεις στον προηγούμενο χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι αυτά μπορούν να ενεργοματοδοτηθούν στα πλαίσια των δύο πρώτων της Ένωσης και Επίσης έχουμε και το άρθρο 311 το οποίο ορίζει ο προπολογισμό χρηματοδότητα στο ακέραιο από ίδιους πόρους. Στην πράξη η πλειονότητα των ε, εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από εθνικές συνεισφορές όπως καλά γνωρίζετε που είναι ποσοστό του ΑΕ και του φόρου προς αξίες επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ρήτρα της ε, γέφυρας που ενσωματώνται, που προβλέπεται τέλο πάντων το άρθρο 48 τη συνθήκη και λέει για την ομοφωνία ε, στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των ιδίων πόρων που αφορά μια συνήθεια νομοθετική διαδικασία για την έγκριση αυτών των πόρων και έτσι το Κοινοβούλιο σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο συμμετέχει, διαμορφώνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι αυτά θέματα τα οποία τα έχουμε διεκδικήσει ε, επανειλημμένα, πολύ σημαντικά. Το σημείο 3 των προτάσεων αφορά Βέβαια θα πρέπει να σεβαστούμε το όριο που έχει τεθεί για την ε, έκταση του κειμένου και εδώ επισημαίνεται η ευκαιρία που παρουσιάζεται από το Brexit, το ώστε να επανεξετάσουμε το σύστημα των μειώσεων και διορθώσεων που είναι αντίθετο με το γράμμα των συνθήκων και μετατοπίζεται έτσι η ουσία των συζητήσεων από την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού στο καθαρό υπόλοιπο για τις συνεισφορές των κρατών μελών. Επίσης, προτείνουμε ότι θα πρέπει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του συστήματος να βασίζεται στην επικουρικότητα και την κατανοησιμότητα από πλευράς πολιτών. Και θεωρούμε επίσης για την κατανοησιμότητα των λόγων της βάσης τέλο πάντων της ε, χρηματοδότησης να υπάρχει σχέση με τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, τους ιδίους πόρους της ε, Ένωσης και συγκεκριμένα έχουμε το θέμα της ενιαίας αγοράς, προστασία περιβάλλοντος, το κλίμα, ενεργειακή ένωση, μείωση ανομοιογένειας προλογικής πολιτικής και αυτά αποτελούσαν και προτάσεις της έκθεσης Μόντι εν τέλει. ότι έχουμε τα πέντε σενάρια για το μέλλον της Ένωσης. Και σχετικά είπαμε ότι θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ακόμα και με κάποιες περικοπές για αυτές τις προτεραιότητες της Ένωσης. Αυτή η χρηματοδότηση θα προέλθει από τους ιδίους πόρους. Αυτές είναι οι προτάσεις που σας ανέφερα μέσα στα μικρά στενά πλαίσια που επιτρέπονται για την έκθεση της ε, γνωμοδότησης. Καλώς και τώρα για το ΕΛΚ. το λόγο Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απολογηθώ που δεν μπόρεσα να παρίσταμε στο, στην πρώτη συνεδρίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ζήτημα αυτό τίθεται επιτάπητος εκ και ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε σε ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και να αναλογιστούμε τα όσα προτείνει η ομάδα υψηλού επίπεδου σε σχέση με τους ίδιους πόρους σε ό,τι αφορά την βελτίωση της λειτουργίας του, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την ε, δουλειά που έκανε, για την γνωμοδότηση που μας παρουσίασε. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να αποστείλει τις ιδέες της στην ε, Επιτροπή του Προϋπολογισμού. Είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να μειωθεί το μερίδιο των εθνικών συνεισφορών. Αυτό θα επέτρεπε να μετακινηθούμε, να απομακρυνθούμε από τις συζητήσεις και να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα και νομιμότητα στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κάποιων δραστηριοτήτων. Αναφέρομαι στο Brexit εδώ συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το ζήτημα των μειώσεων και των διορθώσεων. Τρίτον, χαιρετίζω το γεγονός ότι η γνωμοδότηση αναφέρεται στην ε, υιοθέτηση αποφάσεων σε σχέση με τους ίδιους πόρους. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να αναλογιστούμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις επενδύσεις που γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή θεωρώ ότι οι περιοχές που έχουν ιδιαίτερες προοπτικής σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη ε, ευρωπαϊκή αξία, σε ό,τι αφορά τον τομέα της ανάπτυξης και της έρευνας, αλλά και την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Τέλος, είναι ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον προϋπολογισμό καθένα από αυτά θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ιδέα μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, για παράδειγμα, σενάρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενότητα του προϋπολογισμού, αλλά και να αυξήσουν την πολυπλοκότητα του ζητήματος του προϋπολογισμού. Με όλα αυτά δεδομένα, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συνεισηγητές στις εβδομάδες που ακολουθούν και να μπορέσουμε μαζί να υπογραμμίσουμε τα βασικά ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μόρτε μέσα με τη το VCR. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ την κυρία Μπρέσο για το εξαιρετικό έργο που έχει κάνει. Από ε, ακαδημαϊκή άποψη βέβαια μπορεί να μην είναι αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο το ενόκο ζήτημα, αλλά ε, θα ήθελα εν συντομία να επισημάνω ότι το ECR πράγματι αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο, από διαφορετική οπτική γωνία το ενόκο ζήτημα ε, και θα θέλαμε να κατευθυνθούμε προς ένα ε, ε, ή μάλλον η λογική του ότι μια άμεση με φορολογική βάση η συλλογή φορολογικη βαση συλλογη αυτων των ιδίων πόρων δεν θα ε, μα βοηθούσε σε ό,τι αφορά την περιπλοκότητα του χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη σήμερα δηλαδή οι πολίτε δυσκολεύονται στο να αντιληφθούν πώ ακριβώ νομοθετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε με βάση το πώς ε, μεταφέρονται τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δεν είμαι βέβαιος ότι ένα νέο σύστημα φορολόγησης για την ίσπραξη αυτών των ε, εσόδων θα ήταν κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εμείς θα διταχθούμε σε αυτή την πρόταση. Και επίσης ε, θα διταχθούμε σε αυτή την ρήτρα γέφυρας και η απόφαση με βάση αυτή τη ρήτρα, δηλαδή ναι, οι αποφάσει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα υπόλοιπα ζητήματα, ακριβώ επειδή έχουν τύχθει ε, και με δίκαιο τρόπο, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, αλλά σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα που ανέφερα μόλι τώρα, εμεί διαφωνούμε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Φάβου Καστάλλου. Ευχαριστώ την συνάδελφο πρόεδρε για αυτή την ε, ονομοδότηση που περιέχει πάρα πολλά από αυτά τα σημαντικά στοιχεία και ζητήματα που θα πρέπει να θίξουμε κατά αυτή την προβληματική για του ίδιου πόρου. Βεβαίω και στάθηκε στα θέματα τη ε, επικουρικότητα, τη κατανοησιμότητα του ίδιου πόρου. και θεωρώ επίση όμω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δούμε τι θα γίνει με την συνήθεια θετική διαδικασία από τη μία και την αλλαγή όσον αφορά το σύστημα της ε, ενισχυμένης ειδική πλειοψηφίας. Και όλα αυτά μέσα στην συγκυρία του Brexit, το οποίο νομίζω ότι δημιουργεί συνθήκες ευμενείς για αυτή την ε, κουβέντα. Σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, το σημερινό τοπίο όσον αφορά τις μειώσεις και τις διορθώσεις και βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε το σύνολο της ακτιτομικής του συστήματος όσον αφορά το ότι θα πρέπει να κατησχεί πάντα η αρχή της προστασίας του προϋπολογισμού. Τα συζητήσαμε και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και είπαμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν ε, για να αποδώσει η εργασία μας με την εισηγήτρια και τους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές από ό,τι καταλαβαίνω. δεν Η πρόεδρο αναρωτιέται αν κάποιο θέλει να μιλήσει ω κοιοδή συζητητή ή απλά θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πρόεδρο, λέει ο κύριο Μπάτεν. Είναι ανάγκη λοιπόν να εντοπίσουμε τι βασικέ προτεραιότητε. Γι' αυτό είναι καλό το ότι προς προ αυτήν την κατεύθυνση οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Ε, ποια είναι η, η λογική σε ό,τι αφορά το ποσοστό που δίδεται από κάθε χώρα, το ποσοστό του ΑΕΝ, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Είναι ανάγκη να απλοποιηθεί και είναι ανάγκη οι πολίτες να είναι ενήμεροι. Και συμφωνώ με την παρατήρηση ότι το Brexit είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Αυτό είναι μάλλον ένα δώρο αποχωρισμού από την Βρετανία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τα λόγια του Σίμον Βέιλ. Το 1980 είπε λοιπόν ότι ένα υπεύθυνο κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να α, θεωρεί τον προπολογισμό κάτι δεδομένο, θα πρέπει να κοιτάζει πώς ακριβώς συλλέγεται ούτως ώστε να δει πώς οι συμβολές ε, των εμπλεκόμενων μερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ανάγκη λοιπόν να απομακρυνθούμε από αυτό το πολύπλοκο ζήτημα χρηματοδότησης, ούτως ώστε οι πολίτες να ξέρουν πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνουν, να φορολογούνται άμεσα, ούτως ώστε να μπορούν να καταλάβουν ποιο μέρος των φόρων που πληρώνουν κατευθύνεται προς την χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, ε, θα ήθελα να θίξω κάτι που ανέφερε ε, ο κ. Σπάτεν, ε, το οποίο επί της αρχής ακούγεται ε, πολύ θετικό, καθώς θα έδειχνε στους πολίτες το πόσο μικρό είναι ε, το, το, το ποσοστό των δαπανών που πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το 98% αφορά το εθνικό ή το περιφερειακό επίπεδο των κρατών Μόνο το 2% δηλαδή αφορά τη χρηματοδότηση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο κακή η ιδέα ε, του κ. Πάντων. Ωστόσο, ε, κάτι που θα ήθελα να αναφέρω είναι μια λεπτομέρεια εδώ ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το σχέδιο γνωμοδότηση που μας ε, υπέβαλε εδώ η συγκήτρια, ε, στην πρώτη παράγραφο που αναφέρει ότι αντίκειται και στο γράμμα και στο πνεύμα των συνθήκων. Και στο γράμμα λοιπόν αναφέρεται εδώ και θεωρώ πως δεν είναι σωστό το να λέμε ότι το εφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων ε, αντίκειται στο γράμμα των συνθήκων. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ήταν παράνομο και κατά τη συνέπεια βέβαια θα είχε υπάρξει και δικαστικού χαρακτήρα πλέον ε, την του. Οπότε, αντιλαμβάνομαι ότι ε, αυτό ε, στο οποίο αντιτίθεστε είναι ακριβώ ότι γίνονται αντιληπτοί αυτοί οι διπόροι ω τελικά εθνικέ συνεισφορέ και όχι ω γνήσιοι οι διπόροι. Αλλά όπω είχε αναφέρει και στη δική του έκδοση ο κ. Λεβαντόσκη, πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε με ιδίου πόρου του οποίου επιθυμούμε ως ε, δηλαδή φόρο τελικά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη με βάση ε, το σχετικό επίπεδο ε, ευημερίας τους βασισμένο ακριβώς στο καθάριστο χώριο εισόδημα. Άρα λοιπόν αυτό το προοδευτικό σύστημα φορολόγησης θα πρέπει να προφανώς να εξαρτάται από το σχετικό επίπεδο ευημερίας του κράτους μέλους. Ίσως λοιπόν έχουμε μια επικριτική στάση επειδή εκ πρώτη όψεως δεν δείχνει ακριβώς να αποτελεί ίδιο πόρο ε, και αποτελεί εθνική συνεισφορά, αλλά από την άλλη πλευρά αποτελεί και ένα δικαιότερο τρόπο ίσπραξης ε, αυτών των πόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με κάποιους άλλους, οπότε δεν θα ήμουν ε, απόλυτα αρνητικός σε αυτό το σύστημα που βασίζεται στο ΑΕ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αναφέρουμε αντίκειται στο γράμμα το σύστημα. Ε, ε, φορολόγηση του γράμματος συνθηκών. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρε. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο που θα να πάρει το λόγο, να δώσουμε και πάλι στην ε, μέσα του λόγο. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου, λέει η κυρία Μπρέσο, για τι παρατηρήσει του. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι εύστοχε. βέβαια, έτσι θα βελτιώσουμε τις προτάσεις μας. Και οπότε θα προετοιμαστώ πάνω σε αυτά. Και βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε σε σχέση με τις ε, τροπολογίες. Από ό,τι βλέπω είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος οι γενικές γραμμές. Ε, βέβαια και το Brexit είναι κάτι το αρνητικό για, από πολλές πλευρές. Όμως, εν προκειμένου για μας, μπορεί να μας ε, βοηθήσει ούτως ώστε να απλουστεύσουμε ένα σύστημα το οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο ξεφύγει και εκεί έχουμε όλες αυτές τις ε, εξαιρέσεις, ε, τις μειώσεις ε, και ούτως ώστε να κυριαρχεί τελικά μια σύγχυση για αυτό, μα καλά τα είπε τώρα ο Κόρμπετ. Το σύστημα θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο σε αναλογικότητα όσον αφορά το ΑΕΠ. Και αντίστοιχα λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποίησεις όσον αφορά τη συμμετοχή των χωρών στον προπολογισμό. Εντάξει, το γράμμα της συνεχής προβλέπει τους ε, δύο σπόρους και ακριβώ όπως είπαμε αυτό αφορά πάρα πολύ και και τους ε, πολίτες. Και είναι τελικά η συμμετοχή κάτι σαν ε, δήλωση εισοδήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, έτσι θα πρέπει να γίνεται η συμμετοχή του κόσμου. Έτσι και όχι με άλλους τρόπους. Τέλος πάντων ευχαριστώ όσους μου υπέδειξαν και τόνισαν ότι οι άμεση φόροι πρέπει να αντιστοιχούν στις κοινοτικές αρμοδιότητες όταν αυτοί οι αυτές οι βαρύνσεις Επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το προσέξουμε αυτό. Κατά τα λοιπά, θα μελετήσω τις τροπολογίες και θα τα σκεφτώ όσο γίνεται καλύτερα σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε και θα συζητήσουμε και με τους σκιώδες ηγητές και τελικά θα προσπαθήσουμε να υπάρξει μια ευρεία συνένεση αυτό το θέμα που έχει θεσμικό, συνταγματικό χαρακτήρα γιατί περί αυτού πρόκειται και αυτό είναι και αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε πολύ την Mercedes, λέει ο Θέλω τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα πρέπει να στείλετε τις τροπολογίες σας, ώστε στις 28 να μπορέσουμε να συζητήσουμε και στις 11 Οκτωβρίου, ούτως ώστε να έχουν χρόνο οι συγητές. Και αν δεν υπάρχει αντίρρηση από τους συγητές, μπορούμε να κλείσουμε το ζήτημα αυτό, να περάσουμε στο σημείο 2 της ατζέντα μας που αφορά τις ανακοινώσεις της Προεδρίας και εδώ να σας πω ότι αλλάξαμε την ημερομηνία λήξης για τις ε, τροπολογίες ό,τι αφορά το πολιετές χρήματο ε, δημοσιονομικό πλάνο για τις 15 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Αυτή είναι λοιπόν η ανακοίνωσή μου. Θέλω να περάσουμε τώρα στο σημείο 3 που αφορά τις ανακοινώσεις μου για την τελευταία συνάντηση που είχαμε στις 13 Ιουλίου. Τα παρακάτω ζητήματα συζητήθηκαν και οι συντονιστές προτείνουν. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία, σχετικά με το ψήφισμα της 17ης Μαΐου του 2017, βασιζόμενο στους κανονισμούς 52 και 83 και τους κανονισμούς λειτουργίας. Ο εισηγητές, η εισηγήτρια με συγχωρείτε είναι η Μάιτε Παγκαζαουρτούντου Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση ΑΦΕΤΣΕΝΤΕ για το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ο εισηγητής είναι από το ΕΠΠ, ο Εστεβάν Γκοζάλες Πόνς. Συντονιστές, οι συντονιστές επίσης αποφάσισαν να αντιταχθούν στο, στην ε, ανάθεση της Οίκονος Αρμόδια Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του άρθρου 22 η σύσταση αυτή προβλέπει την αναθεώρηση του πρωτοκόλου 4 που είναι ένα βασικό σημείο των συνθήκων. Η ΑΦΚΟ λοιπόν είναι η αρμόδια επιτροπή, είμαστε αρμόδιοι για τις αναθεωρήσεις των συνθήκων και αυτό θα είναι μια διαδικασία που μάλλον θα είναι δύσκολη. Η πρόεδρος έχει αναλάβει και το ρόλο του εισηγητή. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν υιοθετημένες. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν έγκριση από το γραφείο του Προεδρείου για μια αποστολή στο Ελσίνκι και στην Ρήγα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού ECI. Στη συνέχεια επίσης συζητήσαμε την διαδικασία αναθεώρησης των κανονισμών α, δεν είναι μόνο ένα τα ζητήματα. Ό,τι προταθεί τώρα από την Επιτροπή μας θα αφορά στην αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας. Οι συντονιστές αποφάσισαν να συναντηθούν, να συναντηθούν για να μπορέσουν να συζητήσουν εκτενώς όλα τα ζητήματα αυτά σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς διαδικασιών. Μπορεί να θυμάστε, το Δεκέμβριο του 2016 είχε συζητηθεί το ζήτημα σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς, τις εσωτερικές διαδικασίες για τον προϋπολογισμό, αλλά και τα ανώτατα όρια, για παράδειγμα συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν σε συγκεκριμένα επιδόματα η ομάδα εργασίας πίστευω να μπορέσει να συναντηθεί άμεσα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το ζήτημα αυτό αφορά και την Επιτροπή του Προϋπολογισμού. Το προ, η προηγούμενη συνάντηση που είχαμε στις 20 Ιουνίου, οι συντονιστές συμφώνησαν στην προετοιμασία μιας σειράς εγγράφων εργασίας για το μέλλον της Ευρώπης και τα έγγραφα αυτά εργασίας διανεμήθηκαν στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά το... Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πλαίσιο στην Σπινέλη από τον EPP ο Γιώργη Σόπλεν θα εργαστεί σε ένα έγγραφο με τον τίτλο «Παγκοσμιοποίηση» με τη συνεργασία του ΑΛΤΕ. Από το επίπεδο ο Μάρκους Πίπερ και η Mercedes Πρέσο από το S&D θα δουλέψει πάνω στον εγγραφό EMU, ο Πάολο Ράντζελ από το ΕΠΠ και ο Γιώ Ράινεν από τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Θα δουλέψουν πάνω στον εγγραφό για την άμυνα, ο Έλμαν Μπρόκ από το ΕΠΠ και ο Ραμόν Χαουρέγγι από τους Σοσιαλδημοκράτε θα δουλέψουν πάνω στο έγγραφο EU Finances, η Μαΐτε από το ALDE θα δουλέψει σε ένα έγγραφο που αφορά το citizenship, η Θαγένια Από το ECR θα είναι το άτομο που θα δουλέψει στο έγγραφο Structure and Working Method of the Council με την Κλάουδια Τάπαρντελ και ο Πασκάλ Ντουράντ από τους Πράσινους θα είναι το άτομο που θα δουλεύσει στο έγγραφο Multi-Speed Integration. Έχουμε μια, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία των εγγράφων αυτών. Θεωρούμε ότι τα έγγραφα μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι έτοιμα, θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να καταστήσω σαφές ότι επικεντρωνόμαστε μόνο σε συνταγματικά και σε θεσμικά ζητήματα των πολιτικών αυτών. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Και μόλις μπορέσουμε να συζητήσουμε τα έγγραφα αυτά, θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αναφορές ό,τι αφορά την εφαρμογή, οτιδήποτε θα προκύψει από επιπλέον συζήτηση. Στο σημείο 4 το σήμερα σας διάταξης ε, το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις ε, συνεδριάσεις μας. Ε, η τελική του εκδοχή διανεμήθηκε στις 28 Αυγούστου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρώ πως έχει εγκριθεί. Τώρα, έχετε σχόλια να κάνετε σε σχέση με τα σημεία που κάλυψα. Ε, αντιλαμβάνω πως ο Ρίτσαρντ Κόρμπετ θέλει να σχολιάσει κάτι παρακαλώ. Ναι, σε ό,τι αφορά τα leftovers, τα εναπομείναντα δηλαδή ε, ε, ζητήματα ε, σε ό,τι αφορά το καταστατικό. Ναι, ε, πράγματι συνάντησα όπως γνωρίζετε ε, τον Πρόεδρο και τους ηγητές της, ομάδας, της Επιτροπής Προπολογισμών και αναφερθήκαμε ειδικότερα σε αυτό ακριβώς το, το ζήτημα, δηλαδή της υιοθέτηση κανόνων στο πλαίσιο του καταστατικού του, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Και θεώρησαν λοιπόν ότι ήταν σημαντικό να εγκριθούν αυτέ οι αλλαγέ στο καταστατικό που αφορούν τον προπολογισμό, προτού εγκριθεί επόμενο προπολογισμό, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Έτσι ώστε ο νέο προπολογισμό να εγκριθεί από αυτού του νέου κανόνε. Οπότε ενδεχομένω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό συγκεκριμένο το ζήτημα, δηλαδή τη τροποποίηση των ελόγων κανόνων του καταστατικού, με μια πιο επιταχυμένη διαδικασία από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν ε, την ε, τροποποίηση των κανόνων του καταστατικού. Πρόεδρος. Ναι, ήδη το αναφέραμε αυτό. Ακριβώς ε, για να μην καταστεί όμοιρος εντό εισαγωγικών το ένα ζήτημα από αυτά των υπολείπων ζητημάτων και να μπορέσουμε δηλαδή τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν να τα προωθήσουμε ταχύτερα. Αν δηλαδή στην ομάδα εργασίας γίνεται ήδη μια δουλειά, προφανώς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα ε, κινηθούμε το ταχύτερο δυνατό και να μην υπονομεύσουμε για τα όσα σχεδιάζει να κάνει και η Επιτροπή Προπολογισμών, εκτός βέβαια και αν υπάρχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι που να έχουν αντιρρήσεις, αλλά δεν βλέπουν να ζητάει κανείς το λόγο, οπότε θεωρώ πως μπορούμε να συζητήσουμε αυτή την πρόταση του συναδέλφου ε, Κόρμπετ, ε, η οποία ούτως ή άλλως συζητήθηκε και ήδη ε, συμφωνήθηκε σε επίπεδο των συντονιστών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια σε σχέση με τα σημεία που μόλις κάλυψα. Εάν όχι, να περάσω τόσο σημείο 4 το οποίο ήδη παρουσίασα τη μεσά διάταξη σε ό,τι αφορά λέει, το χρονοδιάγραμμα των ε, συνεδριάσεών μα. Ε, δεν ξέρω αν ζητάει κάποιο ε, το λόγο ή έχει αντιρρήσει, αλλά βέβαια και να είχε κάποιο αντίρρηση δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, γιατί είναι τόσο σφιχτό το χρονοδιάγραμμα που πραγματικά όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τη διαδικασία δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πλέον από την πλευρά μα να τροποποιήσουμε τι ημερομηνίε αυτέ. Οπότε θεωρώ πω εγκρίνεται και αυτό το σημείο και περνάμε στο σημείο 5 τώρα τη ημερησία διάταξη που αφορά στην υιοθέτηση, στην έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Σα ενημερώνω ότι έχουμε εδώ τα πρακτικά τη ε, συνεδρία τη 20 και 21 Μαρτίου, τα οποία ήδη σα έχουμε υποβάλει και εάν πριν από τη λήξη τη σημερινής συνεδρίασης ε, δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση από την πλευρά σα ε, θα θεωρήσουμε εγκεκριμένα και αυτά τα πρακτικά. Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω ότι ο Γκίφερ Χόφστατ, ο οποίο προβλεπόταν να προσέλθει εδώ στην αίθουσά μα στι 5 η ώρα δεν έχει ακόμα καταστάσει. Έχουμε ακόμα 14, 14 λεπτά μέχρι να έρθει. Οπότε ε, στο μεταξύ να σας ενημερώσω σε, σε δύο ζητήματα. Καταρχήν θα γνωρίζετε ότι ε, διαπραγματευόμαστε εδώ και κάποιο καιρό σε ό,τι αφορά το μετρό διαφάνεια το Transparency Register. Δηλαδή, ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 έχει συσταθεί μια ομάδα επαφή στην οποία συμμετέχει και ο Ράινερ Βίλαντ, με δύο κυρίω διαπραγματευτές, η Σιλβή και Γιώμη δηλαδή, που είναι και η πρόεδρος, ε, και εγώ ω δεύτερη, ε, διαπραγματεύτηκα δηλαδή πρόεδρος τη ε, ΑΦΚΟ. Και πριν από το καλοκαίρι είχαμε φτάσει στην οριστικοποίηση τη εντολή, η οποία θα υιοθετηθεί και στο επίπεδο της διάσκεψης των Προέδρων. Και από εκεί και μετά περιμέναμε για σειρά μηνών την εναρκτήνια συνεδρίαση, δηλαδή μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, και αναμένουμε ότι θα λάβει χώρα ε, τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Την ε, Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας. Και ε, εγώ θα σας ενημερώνω τακτικά από τη δική μου πλευρά ως προς την πρόοδο που σημειώνουμε στο πλαίσιο των λόγω διαπραγματεύσεων Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι προβολικά πρόωρο το να αναφέρω οτιδήποτε άλλο πέραν των όσων ήδη ανέφερα και προφανώς η ΑΦΚΟ συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην αλλογοδιαπραγματεύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Brexit, από την πλευρά της ΑΦΚΟ προφανώς πάντως σας ενημερώνω ω προ το τι συμβαίνει μεταξύ των συνεδριάσεων μα, ε, είχαμε ε, συζητήσει επανειλημμένα στο διάμεσο διάστημα με τον Μισελ Μπαρνιέ και ο ε, Γκίβερ Χώστα θα μα ενημερώσει ω προ το τι ακριβώ συμβαίνει στο επίπεδο τη ομάδα καθοδήγηση, του steering group δηλαδή. Ε, τέλη Ιουλίου δηλαδή και αρχέ Αυγούστου έγινε και περαιτέρω συνεδρίαση και από εκεί και μετά εγώ είχα πολλέ συναντήσει. Ειδικότερα δε αξίζει μια συζήτηση που είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας ε, σήμερα και ε, και ε, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής της Κάτω Βουλής, την πρώτη της Επιτροπής της Κάτω Βουλής, τη Χίλαρη Μπέντ, για ε, ε, της Επιτροπής για τα ζητήματα διαπραγμάτευσης του Brexit, για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και μετά έχουμε τις τακτικές ακροάσεις, ας πούμε, έτσι, συνεδριάσεις ε, ε, που θα λάβουν χώρα με, στο επίπεδο της ε, Επιτροπής Καθοδήγησης, αλλά από εκεί και μετά θα μας ενημερώσει σχετικά ο Γκί. Όμως δεν έχει ακόμα προσέλθει, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 5, γιατί είχαμε προβλέψει υπερβολικά πολύ χρόνο για την ομοδότηση συναδέλφου Μπρέσου. Οπότε ας διακόψουμε για 10 λεπτά πάνω κάτω. Αλλά να είστε σα παρακαλώ στην ώρα σα, γιατί πραγματικά πολλά έχουν λάβει χώρα στον διάμεσο διάστημα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει για τον Brexit. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη. Ε, δύο μηνύματα λάβαμε από τον Αιγύη. Το πρώτο ήταν coming, έρχομαι και το δεύτερο είμαι καθοδόν. Αν οπότε ελπίζουμε... Α, κατεύθυνση. Uh, Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, ειδικότερα και εσάς που προσέλθατε ειδικότερα για το συγκεκριμένο σημείο της σημερινής σας διάταξης και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Γκί, να τον ευχαριστήσω για το γνώσο ότι βρίσκεται εδώ μεταξύ μας ε, και για όσους είστε καινούργοι εδώ ε, σε ό,τι αφορά τα αισθήματα ειδικότερα του Brexit, ε, γνωρίζετε καλά το τι συμβαίνει, είναι ο κύριος αρμόδιος ε, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει του Brexit και είναι επικεφαλή ε, τη ομάδα καθοδήγηση του Steering Group ε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώ αυτή ήταν και η ομάδα αρμόδια για αυτέ τι διαπραγματεύσει. Οπότε, α, πάρε το λόγο εκεί με το μικρόφωνο μπροστά σου για να σε καταγράψουμε καλύτερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο, αλλά βρισκόμουν σε μια συνεδρίαση με τον κύριο Μπεντ, ο οποίο είναι ο επικεφαλής της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Κατοπουλής του Ηνωμένου Βασιλείου ε, σε ό,τι αφορά το Brexit. Ενδεχομένω ε, θα έπρεπε να τον προσκαλέσω στην επόμενη συνεδρίαση τη ΑΦΚΟ. Όταν δηλαδή θα επισκεφθεί την επόμενη φορά το Κοινοβούλιο. Τώρα, Γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι ε, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε ε, στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή η διάσκεψη των ε, Προέδρων από κοινού με την Πρόεδρο εδώ της Επιτροπής ΑΦΚΟ που δίνει το στίγμα, θέλετε, την καθοδήγηση για τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρακολουθεί ακριβώ το τι συμβαίνει σε σχέση με το Brexit είναι η ομάδα καθοδήγηση, ο steering group. Ενώ ε, στο ε, ε, Συμβούλιο έχουμε το working group, την ομάδα εργασία και έχουν αντιστραφεί λίγο οι ρόλοι. Δηλαδή συνήθω εμεί έχουμε τι ομάδε εργασία και εκείνοι έχουν την ομάδα καθοδήγηση. Τώρα έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Άρα λοιπόν η ομάδα καθοδήγηση σε συνεργασία με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΑΦΚΟ συναποτελείται από τα μέλη εκείνα τα οποία προφανώς έχουν υιοθετήσει και εκείνα και αποδεχτεί την εντολή η οποία θετήθηκε από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις. Και από εκεί και μετά τα περαιτέρω ψηφίσματα τα οποία θα υιοθετηθούν στο εγγύς μέλλον οι ε, επιτροπέ οι οποίε θα τα υιοθετήσουν θα προσκληθούν και εκείνε προφανώ να συμμετάσχουν στην ε, ομάδα καθοδήγηση. Γιατί τέθηκαν κάποια ερωτήματα από συναδέλφους σας. πώ δηλαδή δημιούργησε η διάσκεψη των Προέδρων αυτή την ομάδα καθοδήγηση και με ποιο σκεπτικό, ποια συλλογιστική. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση που σα δίνω. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχή. Τώρα, ε, στο εντωμεταξύ όπως γνωρίζετε έχουμε τρεις διαπραγματευτικούς γύρου μεταξύ Ένωση, ε, και στιγμή δηλαδή εκπροσώπου τη Ένωση του κ. Μπανιέ και αφετέρου με του εκπροσώπου τη ε, βρετανική κυβέρνηση, υπό την εποπτεία είπαμε εδώ πάντοτε αυτέ οι διαπραγματεύσει τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου και τη ομάδα Κατοδίκηση του Κοινοβουλίου. Ε, στο πρώτο γύρο διαπραγμάτευσης είχαμε καταρχήν απλά την επίσημη έναξη της διαπραγμάτευσης ενώ στο δεύτερο γύρο τον Ιούλιο παρουσιάστηκαν οι θέσει των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τα κύρια ζητήματα προ διαπραγμάτευση. Ο τρίτο ε, γύρο διαπραγμάτευση ήταν ο γύρο τη αποσαφήνιση των διευκρινήσεων ε, μετά δηλαδή από την παρουσίαση. Και ελπίζω πω ο τέταρτο γύρο θα είναι πραγματικό γύρο διαπραγμάτευση, γιατί αυτό είναι και ο στόχο τη διαδικασία. Όπω ε, ήδη ξεκίνησε ε, από την περασμένη εβδομάδα. Ε, όπως γνωρίζετε, η θέση της ε, Ένωσης είναι ότι προτού συζητήσουμε τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου, μια σχέση μελλοντική, η οποία θα πρέπει να είναι σημαντική, να είναι εις βάθος σχέση και προνομιακή μεταξύ πάντοτε Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτού λοιπόν συζητήσουμε αυτή τη σχέση θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε τα της συμφωνίας αποχώρησης ε, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 30 της ε, συνθήκης. Αυτή η συμφωνία λοιπόν σε ό,τι αφορά την αποχώρηση έχει, περιλαμβάνει μία σειρά από σημαντικά στοιχεία ε, καταρχήν ε, σε ό,τι αφορά την ε, κατοχήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών και εδώ αναφέρομαι και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στους πολίτες, Βρετανούς πολίτες οι οποίοι διαμένουν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο τώρα θεματικό πεδίο αν θέλετε είναι η, ε, οικονομική, χρηματική αποζημίωση του διαζυγίου των εισαγωγικών μεταξύ ε, Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τρίτο ζήτημα είναι το ζήτημα των συνόρων. Εξωτερικά δηλαδή σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα νέα εξωτερικά ε, σύνορα ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα ε, των σύνορων εκεί με την Βόρεια Ιρλανδία. Και όπως γνωρίζετε δεν θέλουμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξουν πιο σκληρά εισαγωγικών σύνορων, πιο αυστηρή δηλαδή έλεγχη στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδία, τη Μεγάλη και Ιρλανδία. Και από εκεί και μετά υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα όπω για παράδειγμα τα τη Ευρατόμ, στα οποία δεν θα επισέλθω τώρα, αλλά αποτελούν και αυτά ζητήματα επί των οποίων έχουν εκδοθεί και ε, έγγραφα θέσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά, από την του και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συντάξει αντίστοιχα ε, έγγραφα θέσεις. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα βασικά στοιχεία ε, της Συμφωνίας για την αποχώρηση. Και είχαμε πει ευθύ εξ αρχή ότι εφόσον επιτευχθεί επαρκή πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτά τέσσερα ζητήματα, τότε θα μπορέσουμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης, δηλαδή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση επί της μελλοντικής σχέσης μεταξύ Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου. Τώρα, το ζήτημα του κατά πόσο θα, ποιος θα κρίνει δηλαδή το εάν έχει επιτευχθεί σε πρόοδος ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Ε, είχε προβλεφθεί ε, να γίνει κάτι τέτοιο, ε, δηλαδή να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Εκεί δηλαδή το σκεπτικό ήταν ε, το Κοινοβούλιο από την πλευρά του να θετήσει ένα ψήφισμα αξιολόγησης του κατά πόσο ακριβώς έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα και αυτή ήταν η δική μας πρόταση, δηλαδή το Κοινοβούλιο μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες να υιοθετήσει ψήφισμα το οποίο θα αξιολογεί το κατά πόσο έχει επιτευχθεί ή όχι επαρκή σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου να μπορέσει πλέον να περάσει στη δεύτερη φάση τη διαπραγμάτευση, δηλαδή συζήτηση επί τη ε, μελλοντική σχέση Ένωση ε, και Ενωμένου Βασιλείου. Ή, σε διαφορετική περίπτωση, όπου έχουμε αρνητική αξιολόγηση, μέσα στι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου ε, μήνε να συνεχίσει τι συζητήσει σε ό,τι αφορά την Συμφωνία τη Αποχώρηση. Μετά από την ενημέρωση τώρα που είχα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και σήμερα από τον κύριο Μπαρνιέ, εκείνο που ακούμε είναι ότι είναι πολύ σαφές. Δεν έχει επιτευχθεί επαρτήση πρόοδος ε, σήμερα που να μας επιτρέψει να περάσουμε στη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης. Και Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ στα επιμένου ζητήματα αυτή τη διαπραγματεύση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Θα είδατε ότι δημοσίευθηκε και από τις δύο ε, πλευρές ένα συγκριτικό έγγραφο που απαριθμεί τα επιμέρους στοιχεία αυτών των δικαιωμάτων δηλαδή των ε, πολιτών από τις δύο πλευρές και το οποίο έγγραφο ε, διευκρινίζει το κατά πόσο υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία μεταξύ των ε, δύο πλευρών. Δηλαδή πράσινο χρώμα για τα ζητήματα επί των οποίων υπάρχει συμφωνία και ε, κόκκινο χρώμα για διαφωνία. Χωρί βέβαια να έγινε κάποια συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει πράσινο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα από εκεί και μετά για τα ζητήματα επί των οποίων χρειάζονται περαιτέρω ε, διευκρινήσει. Τώρα, τι κάναμε εμεί με βάση αυτόν τον συγκριτικό πίνακα. Συγκεντρώσαμε από τις διάφορες ε, επιτροπές, τους προέδρους δηλαδή των επιτροπών που συμμετέχουν εδώ ε, και από τους εκπροσώπους της ομάδας καθοδήγησης για το Brexit τα σχετικά σχόλια. Και έλαβα και σχόλια από την ομάδα ECR πάντοτε σε σχέση με αυτό το συγκριτικό πίνακα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς, συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα σχόλια και αύριο το πρωί θα δημοσιεύσουμε στον ιστότοπο τη Ομάδα καθοδήγηση για το Brexit αυτό ακριβώς το έγγραφο, αυτό τον ε, πίνακα, ο οποίος, όπως είπα, αναφέρει στη μία στήλη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωση στην επόμενη της, ε, τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και από εκεί και μετά το αν υπάρχει συμφωνία διαφωνία και τα σχόλια από την πλευρά ε, του ε, Κοινοβουλίου και βέβαια Γιούρι, Λίμπε, Έμπλο, ε, Αύκο και εκπρόσωποι της ομάδας καθοδήγησης είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συντάξει και έχουν συνεισφέρει σε αυτά τα σχόλια που θα περιλαμβάνονται εκεί και βέβαια και τα σχόλια της ομάδας ΕΣΙΑ όπως σας είπα. Αύριο λοιπόν θα δημοσιευθεί αυτό το έγγραφο με αυτό το πίνακα ως επισκόπηση του πού βρισκόμαστε, σε ποια σημεία δηλαδή βρισκόμαστε σε συμφωνία, σε ποια βρισκόμαστε σε διαφωνία και μάλιστα σε διαφωνία όχι μόνο μεταξύ ημών και της ε, Βρετανικής πλευράς αλλά και μεταξύ μόνο των ίδιων, δηλαδή σε ό,τι αφορά δύο συγκεκριμένα ζητήματα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, ε, ε, τι έχει γίνει σε επίπεδο διαπραγματεύση ε, για τα δικαιώματα των πολιτών μέχρι στιγμή, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση των μετακινούμενων συνολικών εργαζόμενων, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ζήτηματα ιατρικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη, να πούμε ότι ναι υπήρξε κάποια πρόοδο ε, στο πλαίσιο των ε, τριών πρώτων διαπραγματευτικών γύρων. Όμω εκείνο το οποίο παραμένει βασικό πρόβλημα για μα με βάση την πρόταση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών που επέβαλε η Βρετανική πλευρά ε, δεν είναι το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών γιατί η πρόταση που κάνει η Βρετανική ε, κυβέρνηση ε, προβλέπει ένα ε, καθεστώς μόνιμα εγκατεστημένου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο προβλέπει πάνω κάτω τα ίδια δικαιώματα με τους Βρετανούς πολίτες πέραν, εκτός από ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση γιατί εκεί εδώ τα ζητήματα μετακατάσταση μια οικογένεια είναι πολύ πιο περιορισμένα. Άρα, όλα αυτά δεν είναι το βασικό μα πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι θα έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο θα συμπεριληφθεί στην Βρετανική νομοθεσία και με βάση το οποίο για να λάβει κανείς αυτή την, το καθεστώς του μόνιμα διαμένοντος ε, θα πρέπει να προβλεί προβεί σε, ένα σχετικό, σε μια σχετική αίτηση και θα κληθεί να τεκμηριώσει, να αποδείξει μια σειρά από στοιχεία, προκειμένου στη συνέχεια η Βρετανική κυβέρνηση να αποφασίσει κατά πόσο θα του χορηγήσει αυτό το καθεστώ ε, το μόνιμα διαμένοντο. Και μάλιστα αυτή η αίτηση δεν θα γίνεται ε, οικογενειακά, θα γίνεται ατομικά. Εάν έχουμε δηλαδή έναν. Ε, έχουμε ο ίδιος ε, σύζυγο και τρία ε, τέκνα θα πρέπει πέντε διαφορετικέ αιτήσει να υποβληθούν από τα μέλη αυτή τη οικογένεια. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμεί σήμερα. Δεν είναι δηλαδή ε, το πρόβλημά μα τα ίδια τα δικαιώματα τα οποία καλύπτει αυτή η πρόταση τη Βρετανική πλευρά σε ό,τι αφορά το καθεστώ του και ούτω ή άλλω το ζήτημα τη οικογενειακή επανένωσης, ε, ε, το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, αλλά το πρόβλημά μας είναι το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό το ζήτημα, ότι δηλαδή θα πρέπει κανείς ο ίδιος να υποβάλει αίτηση και θα ε, κληθεί να αποδείξει ότι πληρεί μια σειρά από προϋποθέσεις. Και το γεγονός βέβαια ότι θα πρέπει αυτή η αίτηση να γίνεται μεμονωμένα, ατομικά από κάθε ενδιαφερόμενο. Ε, δεν ε, θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να γίνει μια τέτοια αντιμετώπιση. Θα πρέπει να πούμε ότι όσοι ήδη διαμένουν μόνιμα στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσουν να χαίρουν αυτών των δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει δηλαδή ε, να τους δημιουργήσουμε, τους επιβαρύνουμε περαιτέρω διοικητικό άκτο ή να πρέπει να τεκμηριώσουν εκ νέου ε, αυτή την μόνιμη διαμονή τους. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για τους Βρετανούς ε, πολίτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου με βάση δηλαδή το ψήφισμα το οποίο εθετήσαμε και το οποίο συγκέντρωσε και συντριπτική πλειοψηφία των ψηφών ότι δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα για τους Βρετανούς ε, πολίτες οι οποίοι διαμένουν ε, στι ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λοιπόν ένα από τα πράγματα που έχουμε πει ω Κοινοβούλιο είναι ότι εάν κανεί διαμένει σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρείται κανονικά διαμένων και μετά δηλαδή από την αποχώρηση της Βρετανίας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να μετακινηθεί κανονικά σε άλλο κράτος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εντάξει, ακόμα αυτή βέβαια δεν είναι η θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Και ε, θα πρέπει να είναι δυνατό και για τους ε, πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες που δεν στη Βρετανία ή Βρετανού πολίτε που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν το, ε, το, το, δικαίωμα να συμμετέχουν στι διάφορε ε, ε δημοτικέ και τοπικέ εκλογέ. Γιατί εδώ δεν τίθεται ζήτημα επικότητα, ε, τίθεται ζήτημα διαμονή σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Και εάν κανεί διαμένει σε μια κοινότητα, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ψήφου στι σχετικέ τοπικέ εκλογέ. Άρα λοιπόν αυτό είναι και αυτό είναι ακόμα ζήτημα ε, επί του οποίου και εμείς ασκούμε πιέσεις για να γίνει δεκτό ε, και αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών, έχει σημειωθεί μια σχετική πρόοδος σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, σε, σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Τίνουμε να συμφωνούμε το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών εξακολουθεί να είναι το γεγονός του πώς θα διευθετηθούν τα ζητήματα που θα προκύψουν σε μεμονωμένη βάση, κατά άτομο. Εμείς από την πλευρά μας, από την ευρωπαϊκή πλευρά και κυρίως από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη προοπτική χωρίς να επιφορτωθούμε με επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, υπήρξε, πρόκυψε το ζήτημα ενός γράμματος που εστάλησε 100 πολίτες Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λέγοντας ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα. Βέβαια αυτό αναγνωρίστηκε ως λάθος, το γράμμα αυτό. ίσως και κάποιοι από τους ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παραπονεθούν για τις επιπλέον ε, διαδικασίες που θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν σε ό,τι αφορά την παραμονή τους ή άλλα έγγραφα που ενδεχομένω να χρειάζονται. Είναι σαφές εν ολίγης ότι για τους πολίτες που ζουν, για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και για Βρετανούς πολίτες που ζουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα γίνονται προοδευτικά όλο και πιο δύσκολα Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό, διότι τα νέα δεδομένα θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι τότε το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προβλέπει τουλάχιστον η τρέχουσα νομοθεσία και οι κανονισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται και δεν θα πρέπει να τους αλλάζουμε γιατί συζητάμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάλι ε, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να εκφραστώ και για τις δύο πλευρές. Και εμείς έχουμε λάβει γράμματα αρκετών ε, πολιτών που παραπονιούνται για, την, για το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το δεύτερο ζήτημα τώρα που θέλω να θίξω και να σας πω πού βρισκόμαστε αφορά την Ιρλανδία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από τους ε, διαπραγματευτές, έχουν σημειώσει προόδους σε ό,τι αφορά τον, την ε, ζώνη ελεύθερης μετακίνησης. Και επίσης σε ό,τι αφορά την... το βασικό ζήτημα των συνόρων, το οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε επιπλέον και από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια αποδεκτή λύση και από τις δύο πλευρές, ό,τι αφορά το ζήτημα των σύνορων και πάλι. Αλλά και σε αυτό το γενικότερο ζήτημα του αόρατου συνόρου. Έχω αστιευτεί λίγο για αυτά τα αόρατα σύνορα. Έρχομαι από μια χώρα που ο σουρεαλισμός κάτι σημαίνει αν έχετε στο μυαλό σας πίνακες του Μαγκρίτ. Αυτό δεν είναι μία πίπα, σε πάζιν πίπα. Όταν κοιτάζω λοιπόν τον πίνακα αυτό ή όταν α, ε, αναλογίζω με τις συζητήσεις αυτές για το αόρατο σύνορο, σκέφτομαι το Μαγκρίτ και όλα αυτά τα αόρατα σύνορα. Αυτό είναι ένα σύνορο ή δεν είναι ένα σύνορο. Μπορώ όμως να φανταστώ ότι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό το ζήτημα του αόρατου συνόρου. Πληρώνεις με ένα νόμισμα από τη μία πλευρά του συνόρου και με ένα άλλο από την άλλη πλευρά του συνόρου. Και μια σειρά από πράγματα διαφέρουν στην Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία, σε ό,τι αφορά το νομικό τους πλαίσιο, για παράδειγμα, το νομικό του σύστημα. Αλλά και τα όρια ταχύτητας, όπως λέει ο κύριος Κόρμπετ. Είναι σαφές όμως ότι αυτό που εμείς ψάχνουμε ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι η, επιπλέον ε, ενδυνάμωση του συνόρου αυτού. Θέλουμε ένα σύστημα που να είναι καλό όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για αυτούς που ε, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και από αυτό προκύπτει το ερώτημα, τι, τι είναι αυτό το σύνορο λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη συζητάμε μελλοντικέ σχέσεις. Γιατί αν για τον έναν ή τον άλλο λόγο η Βρετανία εξακολουθεί να είναι μέλος της Θελωνιακής Ένωσης, για παράδειγμα, ε, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό όμω δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο που μα αφορά είναι πού ακριβώ θα βρίσκεται το σύνορο και πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα πιο ισχυρό σύνορο σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, γιατί και οι δύο πλευρέ, τόσο η Ιρλανδική Δημοκρατία όσο και, το βόρει, όσο η Βόρεια Ιρλανδία, έχουν συμφέρον να επιληθεί το ζήτημα αυτό και πώς θα μπορέσουμε να, να πραγματοποιούμε ελέγχου για παράδειγμα Υπάρχουν περισσότερα από 260 σημεία, όπως με ενημέρωσε ε, ο Ιρλανδός Υπουργό μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας. 260 σημεία ελέγχου. Μήπως είναι μόνο τα, τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο τα σημεία που θα πρέπει να παραμείνουν ως σημεία ελέγχου. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που ήθελα να δείξω. Το τρίτο έχει να κάνει με τον οικονομικό συμβιβασμό. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος σε ό,τι αφορά τις οικονομικές αποζημιώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων έθεσε σε αμφισβήτηση την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για τη θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την, ε, την ε, απέτηση δηλαδή για οικονομική αποζημίωση. Θεωρώ ότι πιστεύω σε μια συνέντευξη τύπου συζητήθηκε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις αλλά όχι νομικές υποχρεώσεις. Εμείς από πλευράς μας στο ψήφισμά μας είπαμε ότι πέρα από το 2019 μπορεί και να προκύψουν οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι και το αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που είχαν αναλυφθεί πριν το 2019. Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ μιας δέσμευσης και αποπληρωμής. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα που, που έλαβα στην πράξη, γιατί εγώ ήμουν δικηγόρος. Όταν λοιπόν ανέλαβα τη θέση του Υπουργού Οικονομικών ε, ήταν λίγο πρόβλημα αυτό για μένα. Το να μπορέσω να, μάθω όλα αυτά τα πράγματα που μου χρειάζονταν. Δεν ήταν ιδιαίτερο προσόν το πτυχίο τη νομική. Κατάλαβα όμω τη διαφορά ανάμεσα σε μια αποπληρωμή και μια δέσμευση. Δεν μπορεί λοιπόν να πει ότι μέχρι από το 2019 και μετά δεν πληρώνουμε τίποτα, γιατί μπορεί να έχουμε αναλάβει μια σειρά αποδεσμεύσει, οι οποίες να είναι δυνατόν να αποπληρωθούν μετά την αποχώρηση, μετά το 2019. Ή μπορεί να προκύψουν ε, επιπλέον υποχρεώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους να παράγουν την ανάγκη αποπληρωμής. Και αυτό δεν το γνωρίζουμε σήμερα, πώς ε, θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε πώς θα προκύψει μια ε, επένδυση που έχει γίνει τώρα. Αν υπάρχει μια εγγύηση για την επένδυση αυτή, δεν ξέρουμε αν η επένδυση θα είναι επιτυχής και η εγγύηση δεν θα χρειαστεί να χρηματοθεί. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα ε, πρέπει να, να συζητηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Είναι ανάγκη να τα αναγνωρίσουν και οι δύο πλευρές ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα του οικονομικού συμβιβασμού. Και εκεί η πρόοδο είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Και τώρα για να δούμε. Τι θα γίνει στου επόμενου ε, γύρου. Μάλλον στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων θα πάμε την ε, τέταρτη και όχι την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και γιατί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση της ε, Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Προβλέπεται για τις 21 Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν θα ήταν σωστό να μπλεχτεί αυτή η παρέμβαση με τις διαπραγματεύσεις. Άρα μάλλον, μάλλον αυτός ο γύρος θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Επίσης, Θα προτείνω στην διάσκεψη των ε, Προέδρων σήμερα να υπάρξει ένα νέο ψήφισμα από την Ολομέλεια για την πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου, 3 με 4 Οκτωβρίου, για τις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά στοιχεία, τα δικαιώματα των πολιτών που βρισκόμαστε, τι θέλει το Κοινοβούλιο για το πόσο έχει το, το θέμα Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία και επίσης για την πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων. Και μετά πάμε για τον πέμπτο γύρο. Τώρα βρισκόμαστε στον τέταρτο, είπαμε. Άρα λέμε για την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και τότε θα έχουμε τον ε, πέμπτο γύρο τον Οκτώβριο. Θεωρώ δε ότι πριν στο Συμβούλιο θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί αξιολόγηση του πώς, ε, πώς έχουν τα πράγματα, σε ποιο σημείο βρίσκονται και οπότε πάμε για αυτό τον κρίσιμο πέμπτο γύρο πριν το Συμβούλιο όπου και θα γίνει αξία αξιολόγηση τον Οκτώβριο. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι σωστή κίνηση από το Κοινοβουλίο να αξιολογήσει το τι γίνεται με τους πολίτες, ε, τι γίνεται με τα χρήματα οικονομικά, ε, γενικά πώς προχωράμε για τα θέματα του συνόρου Ιρλανδίας, Βορειοϊρλανδίας σε ένα τέτοιο ψήφισμα το οποίο θα κατέβει τέλη Σεπτεμβρίου το συζητήσουν πολιτικές ομάδες και μετά να πάει στην Ολομέλεια. 3 ή 4 Οκτωβρίου. Και ανάλογα με το τι θα κρίνει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Αυτά, Πρόεδρε, αυτό το τοπίο μπορώ να σας περιγράψω. Και ευχαριστώ να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις από τους ε, συναδέλφους. Γεια σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εξαντλητική σου παρουσίαση και τώρα να δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους. Πρώτα πρώτα η Μαρτίνα Άντερσον. Είστε Να σε ευχαριστήσουμε εκεί μία ακόμη φορά για την παρουσίασή σου. Πίστευω ότι για πολλούς από εμά εδώ στο Κοινοβούλιο αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο μέρα με την ημέρα τις επιπλοκές που θα έχει αποχώρηση αυτή και το γεγονός ότι υπάρχουν παραπάνω από 300 συνοριακά σημεία. Και οι επιπλοκές είναι δύσκολο να επιληθούν. Δεν έχουμε καταφέρει να τις λύσουμε εδώ και 100 χρόνια. Και το γεγονός ότι θεωρείται προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά εμείς στην Ιρλανδία. Χαιρόμαστε που η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής Good Friday Agreement είναι κάτι το οποίο συζητείται, είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται. Βεβαίως μας ανησύχησε η ανάγνωση του υπόλοιπου εγγράφου, γιατί δεν θέλουμε να μας παρηγορήσετε δεν θέλουμε να μας πείτε ότι δεν χρειάζεται σύνορο, αλλά μετά να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο το σύνορο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει αν αόρατο σύνολο. Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μια τεχνική λύση Μαθαίνουμε τώρα ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα αυτό. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτεί η εν λόγω συμφωνία από το Κοινοβούλιο και από την Καμισιόν, από την η συμφωνία Good Friday. Αν ρίξετε μια ματιά στις νομοθετικές πράξεις που θέτουν σε λειτουργία τη συμφωνία αυτή του 1998, είναι σαφές ότι οι υπουργοί δεν μπορούν να παράξουν νομοθεσία που να μην είναι συμβατή με τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνος τρόπος που το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να προστατέψουν την εν λόγω συμφωνία στο σύνολό της είναι να εξασφαλίσουν ότι με τη συμφωνία αποχώρησης η συμφωνία Good Friday θα παραμείνει ενισχύ. Θεωρώ επίση, σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση του συνόρου, εκτός και αν μπορέσουμε να έχουμε το νησί στο σύνολό του στην Τελωνιακή Ένωση, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πώς γίνεται δηλαδή να έχεις ένα κομμάτι της Ιρλανδίας ως μέλλον της, μέλος της Ένωσης και ένα άλλο όχι. Μπορείς να αναλογιστείς οποιοδήποτε πρόγραμμα. Πώς είναι δυνατόν να έχεις διαφορετικούς ρυθμιστικούς κανόνες σε ένα και μοναδικό νησί. Πρέπει μάλλον να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση στο πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε του, τα δικαιώματα των πολιτών. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα προστατευτούν, αλλά τα 1,8 εκατομμύρια πολίτες που βρίσκονται στο βορρά του νησιού, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους θα προστατευτούν. Ματίνα, σε ευχαριστούμε και τώρα πριν δώσουμε το λόγο στους άλλους συναδέλφους. Παρακαλώ να τηρήσετε αυτό το των δύο λεπτών γιατί έχουμε μόλις 40 λεπτά και θέλουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει ερωτήσει από πλευρά του και... Mm, today on what, uh, in contrast, the... Ε, σήμερα, γιατί βλέπετε από την άλλη μεριά εσείς τα θετικά, αλλά τα μίντια στην ε, Αγγλία τα λένε όλα μαύρα και ε, λένε ότι όλα τα διέπει κάτι σαν η εκδίκηση και λοιπά. Καταλαβαίνουμε πού το πάνε, αλλά δεν θέλουμε να σας πούμε ότι εμείς ως εσύ θέλουμε αρνητική θέση, αλλά από αυτά τα 11 σημεία τα οποία έχουν περάσει από διαμεταξύ μέχρι τώρα, από αυτά τα, τα 11 σημεία, μόνο τρία, τρία σημεία παρουσιάζουν πρόβλημα. Άρα, ε, οκτώ σημεία έχουν ε, προχωρήσει. Άρα, τι είναι αυτά που λένε τα, τα, τα και ο κύριο Μπαρνιέ γενικότερα στην κατάστημα σκηνή. Αλλά μα είπατε σε τι γίνεται με αυτά τα τρία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεταξύ των άλλων είναι αυτό το ζήτημα το, το, το χρηματοοικονομικό. Είδα του υπολογισμού και από ό,τι καταλαβαίνω, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει το 19, όπω προβλέπετε, ε, τότε θα προβλέπονται 26,5 δις τα οποία θα πρέπει να δοθούν ως επιστροφή. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η επιστροφή υπολογίζεται σύμφωνα με τη Συμφωνία των Επιστροφών η οποία έκλεισε εδώ και κάτι δεκαετίες. Οπότε το θέμα είναι αυτή η επιστροφή, αυτά τα 26 και μισό δις, ε, πώς θα, θα καταβληθούν. Ξέρετε, ε, είχατε κάποια ενημέρωση και αν όντως προτείνει 26,5 δισεκατομμύρια και από ό,τι ακούσαμε στο Σαββατοκύριακο έχουμε επίσης και ένα ποσό 50 δισεκατομμυρίων το οποίο συζητείτε ε, τότε το ποσό που θα οφείλει το Ηνωμένο θα είναι 20,5 δις. Άρα για πέστε μου, αν μας διαφωτίσετε θα είναι πολύτιμο. Εμείς ευχαριστούμε, Νταϊάν, λέει πρόεδρος. Έχω εγώ τώρα το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και θα σας τα πω και στα Ιταλικά για να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Θεωρώ πάρα πολύ ακριβή τα όσα μας εξήγησε ο Γκίφερ Χόφστατ για αυτά τα θέματα προστριβής διαφωνίας που αφορούν την Συμφωνία Απαχώρησης. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε το θέμα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πέραν των άλλων ε, σημείων που αναφέρατε γιατί νομίζω ότι εδώ ακόμα τα πράγματα είναι τόσο σαφή. Τώρα αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι καταλαβαίνω και ε, θεωρώ ότι θα, πρέπει να γίνει αυτή η αποχώρηση. Οπότε και έχουμε ε, τώρα σε αυτή τη φάση ε, πρόοδο και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην δεύτερη φάση κλπ. Δεν θέλω όμως να μου πείτε. Αναφέρεται στο Μενού Βασίλειο ότι όλο και περισσότερο κατεπήγει τον με μεταβατική συμφωνία, κάποια ενδιάμεση συμφωνία. Δηλαδή, βλέπουμε να υπάρχει ολόνα και μεγάλο συνασπισμό δυναμίου πέρα αυτού στη συνδιάμεση συμφωνία, Οπότε θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η Τελωνική Ένωση, η ενιαία αγορά κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτα, πρώτα, πριν τις οποιασδήποτε συζητήσεις θα κρυφθούν όλα αυτά. Πριν το Ηνωμένο Βασίλειο βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κοινωτικό δίκαιο. Άρα, για πέστε μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την ε, διευθυντική ομάδα της Steering Group, τι γίνεται. Υπάρχει πρόθεση συζήτησης αυτή τη συνδιάμεση συμφωνία πριν, πριν κλείσει η συμφωνία της αποχώρηση Δεύτερον, δεν μιλάμε για αυτή την μεταβατική συμφωνία. Υπάρχει τα Άγγλων να εξαιρούν το θέμα των ε, Ευρωπαίων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή διαλέγουν το ότι θα ε, μπει στη συμφωνία. Τσέρι, Πίκινγκ. Όμως θα πρέπει να κάνουμε και με τη σειρά μας ε, μια περιχαράκωση, μια προστασία της συμφωνίας υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών στην Βρετανία. Και κλείνει το μικρόφωνο να συνεχίζει να μιλάει πρόεδρος. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριος Σέπφλ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μας τα εκθέσατε με τόση πληρότητα το τι ήθελε τις εβδομάδες. Έχω τώρα κάποιες ερωτήσεις και θα πρέπει να σας τα πω τηλεγραφικά πρώτα πρώτα νομίζω ότι αυτό το οποίο αντικρίζουμε είναι το ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος, ποιος, ποιος, ποιος ε, είναι στο τιμόν των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει αμφισβήτηση από πλευρά των ε, Βρετανών, υπάρχει αμφισβήτηση και ε, νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Κατά δεύτερο λόγο δεν πιστεύω από αυτά που διαβάζω ότι αποδέχονται οι Βρετανοί τη διάκριση μεταξύ εντολή σε πλευρά Συμβουλίου και από την άλλη μεριά των ενεργειών του Μπαρνιέ. Νομίζω ότι ε, αυτή είναι η καινούργια θεματική, ότι δηλαδή κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη ευελιξίας. Δεν νομίζω ότι διαβάζουν καν τα έγγραφα από το Συμβούλιο ή από τον Μπαρνιέ. Και να τα διαβάζουν δεν καταλαβαίνουν, έτσι νομίζω. Τώρα, το θέμα είναι η Βρετανική κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ αρνητική, δεν βοηθά καθόλου όσον αφορά το να πάμε προς ε, κάποιο αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Παρά το ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον τους. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η προσέγγιση των Βρετανών είναι το ότι δεν είναι κάτι το δεδομένο, το δικαίωμα του να παραμείνει κανεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει κανεί να αποδείξει, να φέρει ο καθένα το βάρο αποδείξεω του ότι δικαιούται να παραμείνει, να διαμείνει. την άλλη μεριά, κατησχύει γνώμη του Westminster, του Κοινοβουλίου, και άλλο μπορεί να ανατολεί πια από τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο. Τι θα γίνει. Αν όχι σήμερα, ας πούμε ότι σε 10 χρόνια η κυβέρνηση λέει δεν τους στέλνουμε όλους αυτούς τους μετανάστες από την υπηρετική Ευρώπη εδώ. Τέλος. Είπατε τίποτα για την Ελία, έτσι από περίεργεια το λέω. Γιατί αυτό και αυτό θα είναι τα πιο δύσκολα. Τι γίνεται με... Πώς, πώς θα διαχωριστούν τα δανέζικα ψάρια από τα βρετανικά ή από τα βέλγικα. Ναι, ναι, θα είναι απάτριδες, θα είναι ανηθαγενείς αυτά τα ψάρια. Ευχαριστώ και, και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Χόφστατ για αυτή την ενημέρωσή του. Για να είμαι πολύ σαφής, ε, να πω πως ε, ε, οι ομάδες διαπραγμάτευσης και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν πολύ συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές και ακριβώ η ε, κατοχήρωση των δικαιωμάτων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από αυτέ τι κόκκινε γραμμέ. Οπότε αυτό που συζητάμε εμεί εδώ σήμερα είναι το πότε και πώ μπορούμε να ενημερώσουμε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ε, πραγματικά ανησυχούν για το μέλλον του σε σχέση με το καθεστώ που θα ισχύει για αυτού στο μέλλον. θα μπορούσαμε βέβαια να αυξήσουμε την πίεση, γιατί και η Βρετανική πλευρά διαπραγμάτευση θα πρέπει να δώσει τι ίδιε αυτέ απαντήσει στου δικού τη ε, ε, Βρετανού ε, πολίτε. Και αυτό με οδηγεί και στο δεύτερο ζήτημα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αποζημίωση, τι σχετικέ πληρωμέ που θα πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη έχουμε, βρισκόμαστε σε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Και από εκεί και μετά τι θα γίνει από το 2020 και μετά. Δηλαδή η δυνατότητα η δική μας να σχεδιάσουμε τις ε, μελλοντικέ ε, εξελίξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αφορά το 2020 είτε το 2028 εξαρτάται και από αυτά εδώ και νομίζω πως θα γίνει και μια αναφορά ε, και, από τον ε, πρόεδρο τη Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν νομίζω πως η σύνδεση αυτών των δύο ζητημάτων μεταξύ τους αποτελεί τελικά ένα γενικότερο ερώτημα ως προς το εάν υπάρχει τελικά μία ε, στάση, αν θέλετε, αξιόπιστη με από την πλευρά των διαπραγματευτών, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις στους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ε, τον Χέλμου, τώρα ο κύριος ε, Μαντίνας έχει το λόγο. Κυρία Μαγκίνα, η Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Αγγί για αυτή την ενημέρωση. Εάν ε, ε, ρώταγε κανείς ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα από όλα τα σημαντικά ζητήματα. Με βάση την παρουσίαση που μας έκανε ήταν πρώτο το ζήτημα το ε, χρηματονομικό και από εκεί ε, ε, και μετά τα, ε, τα σύνορα και τελευταίο αυτά που αφορούν τους πολίτες. Και εδώ θα συμφωνήσω σχέση με αυτό το ζήτημα με τον James, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο σημαντική η ειρήνη από ότι τα χρήματα. Και πράγματι αυτή τη στιγμή τα σύνορα είναι πραγματικά όρατα εδώ, και Λανδίας. Στη δική μου δηλαδή, στη δική μου περιοχή, στο Ντόνικον, ε, είδα ότι υπάρχουν αυτά τα τα σύνορα. Ε, λόγω των πλημμύρων ταξίδεψα και τέσσερις φορές ε, πέρασα τα σύνορα. Οπότε πραγματικά τίθεται εδώ ένα ερώτημα του πού θα γίνονται οι έλεγχοι, πώς θα αστυνομεύουμε αυτά τα 300 σημεία συνορικής γιατί αφού έχει πλέον ισχύσει ήδη και εφαρμόζεται η Συμφωνία της Παρασκευής, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να επιστρέψουμε σε μια ε, φάση πριν από εκείνο. Οπότε ε, θέλουμε Ε, για να διατηρηθεί η κατάσταση με την Ιρλανδία όσο έχει σήμερα, τότε θα πρέπει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ε, στην νέα Ιστορική αγορά ή στην τελωνιακή ένωση. Ακόμα και αν λάβουμε βέβαια αρνητική απάντηση από την πλευρά του. Γιατί οι πολίτε τη Βορείου Ιρλανδία Ε, υπερψήφισαν, ε, το, το, ε, καταψήφισαν το, το Brexit και ακόμα και εκείνοι που συμφώνησαν με το Brexit είπαν, μου, έχουν μιλήσει μαζί μου και μου είπαν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στη φάση σε ό,τι αφορά τα σύνορα πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, πραγματικά είναι εδώ λεπτό το ζήτημα και η διαδικασία ε, προκειμένου δηλαδή να διασφαλιστεί ή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του κατά πόσο θα μπορέσει η Βόρεια Ελληναδία πράγματι να παραμείνει ε, στην Τελωνιακή Ένωση και στην Εννέα Αγορά προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς σύνορων όσο έχει σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω πολλά ερωτήματα που θέλω να θέσω, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο, οπότε θα θέσω μόνο ένα σε ό,τι αφορά την αποζημίωση από την πλευρά τη ε, Μεγάλη Βρετανία. Ε, αν υπάρχει εδώ πρόβλημα, αυτό οφείλεται ε, στην αναποφασιστικότητα από την πλευρά τη Βρετανική κυβέρνηση. Ουσιαστικά ο κύριο Ντέβι τι είπε. Μηδενικό είναι το ποσό που προτείνουμε αυτή τη στιγμή και α δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Πάντω, νομίζω πω. Ο κύριος Βερχόφστατ είπε ότι δεν υπάρχει νομική βάση σε ό,τι αφορά αυτή την αποζημίωση, αλλά μόνο ηθική υποχρέωση. Η μόνη όμως ηθική υποχρέωση κατά τη δική μου άποψη είναι αυτή που αφορά την καταβολή των μισθών, των συντάξεων και άλλων υπαλλήλων δηλαδή ε, της ε, Επιτροπής ε, και βέβαια από εκεί και μετά έχουμε και τους υπολείπους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πώς συμβάζεται αυτή η ηθική υποχρέωση, αυτό το ποσό με τα 100 εκατομμυρία που ακούσαμε κάποτε και από εκεί και μετά ακούσαμε ότι ε, είναι, θα είναι με καταβολή στο 2020, τελικά πήγαμε στο 2023. Οπότε το ερώτημα που θέτω είναι ποιο είναι τελικά το ποσό που υπολογίζεται και μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί. Ε, από εκεί και μετά, εκείνο που θα έπρεπε να είχε κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτέ τι αναλήψει υποχρεώσεων στον προπολογισμό είναι να, να αντιληφθεί από τότε ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω αναλήψει υποχρεώσεων. Ε, δηλαδή, πάντοτε όταν υπάρχουν λιγότερα έσοδα, λιγότεροι πόροι, τότε όλοι θα πρέπει να μειώσουν σχετικά τι δαπάνε του. εγώ δεν θεωρώ ότι η Βρετανία χρωστάει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και αν σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε αφορούμε μόνο, έχουμε να κάνουμε μόνο με καθαρή συνεισφορά. Δηλαδή, βγάλουμε την ε, έκπτωση και τις σχετικούς περιορισμούς, το συνολικό ποσό από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2020 33,7 δις. Ε, και βέβαια με την καταβολή ε, ποσών κάθε χρόνο μειώνεται αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν μέχρι το 2019 το υπολοιπόμενο ε, ποσό θα είναι 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και μετά βέβαια έχουμε και τις σχετικά rebates, τις εκτόσεις, δηλαδή τις μειώσεις οι οποίες επιβάλλονται ένα χρόνο μετά. Άρα λοιπόν, ακόμα ε, κι αν φύγουμε το 2019, δεν σας οφείλουμε τίποτα ως Μεγάλη Βρετανία. Οπότε, συνοψίζοντα, ποια είναι η νομική βάση επί τη οποία αξιώνεται εδώ την καταβολή αυτού του ποσού. Γιατί δεν περιβλάβεται κάτι στο άρθρο 50 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πείτε μα λοιπόν ποια είναι η νομική βάση και πείτε μα με βάση ε, ποιου υπολογισμού καταλήξατε σε αυτό το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων. Για να καταλάβουμε τελικά και εμεί και η Βρετανική κυβέρνηση τι ακριβώ εννοείται. Ευχαριστούμε. Πραγματικά σα ζητώ να είστε σύντομοι να μην ξεπερνάτε το 1,5 ή 2 λεπτά, γιατί έχουμε τόσους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Περνάμε τώρα στον επόμενο μιλητή. Ο κύριε Μπρέσο, ο κύριος, ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ, έχει το λόγο. Είναι πολλές ε, ερωτήσεις που θέλω να ρωτήσω και ήδη τις ρώτησαν οι συνάδελφοι. Ίσως, Γκί, αν έχεις χρόνο στο τέλος να κάνεις κάποιο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των Βρετανών Υπουργών ε, για τον εκβιασμό, τον υποτεθόμενο εκβιασμό α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η επίρρηψη ευθυνών στι Βρυξέλλε που προσπαθούν να υποφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από την επικείμενη αποχώρηση των Βρετανών. Ευχαριστούμε η Mercedes Πρέζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Και εγώ θεωρώ ότι είναι από τα σημεία από τον οποία νομίζω ως κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε να ξεκαθαριστούν τα πράγματα είναι η διαδικασία, οι λεπτομέρειες του πώς ορίζονται οι συγκρούσεις γιατί ε, είναι το θέμα του πώς θέλει κάθε πλευρά να ρυθμιστούν τα θέματα που αφορούν την δικαιοσύνη. Ε, Βεβαίω και πρέπει να δημιουργηθούν προστρεβές και διαφορές. Ας πούμε, όταν μιλούμε για δικαιώματα των ε, πολιτών, μιλούμε για εκατομμύρια πολιτών και ατομικών δικαιωμάτων. Άρα θα είναι δύσκολο να γίνει η σχετική διαχείριση της πολιτικής για τα σύνορα ή τι θα γίνει με την χρηματοοικονομική ε, συμφωνία που βέβαια όταν ρυθμιστεί θα αφορά μόνο τις ε, δύο πλευρές συνολικά. Άρα θα πρέπει προσεκτικά να ε, προβληματιστούμε όσον αφορά το τι εντολή θα πρέπει να δοθεί όταν περάσουμε στην δεύτερη φάση. Ευχαριστούμε την Mercedes το λόγο έχει ο συναδελφός Σελίμωβιτς. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο και τον Κίβερ για την ενημερωσή του. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι κατά πόσο εσείς κύριε Βερχόφστατ έχετε μία αίσθηση σε ό,τι αφορά την, το, την πιθανή συμφωνία των θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα αναφέρομαι σε υποχρεώσεις, πιθανές υποχρεώσεις, θα έχουμε συγκεκριμένα νούμερα, αλλά υπάρχει κάποια συμφωνία σχετικά με τα ζητήματα που θα πρέπει να αποπληρωθούν. Ποια είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Υπάρχει συμφωνία τουλάχιστον σε αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο έχετε μια αίσθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει την κοινή γνώμη για το κατά πόσο πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία, όποιοι και να είναι οι όροι της συμφωνίας αυτής, θα, κατά πόσο η κοινή γνώμη είναι προετοιμασμένη για το ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια συμφωνία. Για μένα, αν ακούσω την δημόσια συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τι λένε οι συνάδελφοι, στο κοινοβούλιο περισσότερο μου φαίνεται ότι έχουν την αίσθηση ότι είναι ένας ανταγωνισμός, ποιος θα φανεί πιο άμεμπτος δεν υπάρχει αίσθηση ότι πρέπει να βρεθεί ένας κοινό τόπος, γιατί και φτάνουμε στο τρίτο ερώτημά μου. Αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει και τις μελλοντικέ σχέσεις μας. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε μια κάποια σχέση στο μέλλον με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι δεν σας χρωστάμε τίποτα. Οκ, δεν θέλετε λοιπόν να έχετε καμία απολύτω σχέση μαζί μας. Γιατί φαντάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο θέλουν να έχουν μια κάποια οποιαδήποτε σχέση, όπως και να τη φαντάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ακούμε καθόλου χρήματα, καθόλου αποπληρωμή, καμία σχέση. Αυτό μου φαίνεται έτσι κάπως ε, δύσκολο να το καταλάβω. Ποια είναι λοιπόν η δική σας γνώμη πάνω στο ζήτημα αυτό. Ούτω ώστε να μπορέσουμε καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και να έχουμε μια μελλοντική σχέση που να είναι αμοιβαία υπόφελης. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος, ο Μαξ Άντερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Βερχόφστα για αυτήν την ενδελεχή ενημέρωση. Αμέσως μετά το δημοψήφισμα ανησυχούσα ότι κάποιοι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θελήσουν να φερθούν σκληρά στην Βρετανία, ούτω ώστε να αποτρέψουν άλλους από το να αποχωρήσουν. Και αυτό θα μπορούσε να είναι υπερβολικό. Αυτό που βλέπω όμως τώρα από πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι η ανικανότητα των Τόρις καθιστά την κατάσταση πολύ χειρότερη για τη Βρετανία, πολύ χειρότερη από ό,τι κανείς μπορούσε να φανταστεί. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, οι διαπραγματεύσεις κινούνται με έναν ρυθμό που θα μας επιτρέψει να έχουμε μία συμφωνία πριν, την, πριν τη λήξη της περίοδου των δύο ετών που έχουμε θέσει εξ αρχής. Και το δεύτερο ερώτημα, βλέπω ότι η θέση των Βρετανών είναι κάπως αδύναμη. Ευχαριστώ. Έχουμε τους δύο τελευταίους ομιλητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συναδελφό Φερχόφτακ για την εισήγησή του που ήταν τόσο πλήρης. Είχαμε πάρα πολλέ ερωτήσεις, οπότε έχω καλυφθεί βεβαίω και εγώ θεωρώ ότι πάντα τα δικαιώματα των πολιτών είναι κορυφαία προτεραιότητα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ασάφειες όσον αφορά αυτά τα αόρατα σύνορα, αυτό το οποίο το Λονδίνο έχει προτείνει για τη Ιρλανδία ως λύση για τη γενική αίσθηση, είναι το ότι ε, αυτό το οποίο γίνεται είναι κάτι σαν παρτίδα πόκερ. Αυτό το σκεφτούμε, γιατί έτσι πάμε για να λύσουμε τα πιο ακανθόδη. Δεν περιμένω τίποτα ε, ε, κεραυνοβόλες πρόοδους στις αμέσως επόμενες φάσεις έχω να σας πω από ό,τι άκουσα και από του συναδέλφου ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτή την κοινή δήλωση Ιαπωνία και ΙΠΑ ε, γιατί ο Σινσουάμπε και η ΜΕΙ επίσης τοποθετήθηκαν όμως αν είναι και όσο είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς η Τερέζα ΜΕΙ προβαίνει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις διμερεί. όμως αυτό το είπαν, υπήρξε πολιτική βούληση ε, και η Ιαπωνία βεβαίω και αυτή περιμένει να δει πώ θα ωφεληθεί από τον Brexit, αλλά εγώ περιμένω να δω τι θα κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και αυτό το θέμα όπω και άλλα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στι διαπραγματεύσει και θα πρέπει και εκεί να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και να δούμε τι εναλλακτική υπάρχει. Πώς μπορεί κάποιος ο έτσι να κάνει τέτοιες διαπραγματεύσεις. Γιατί όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, αυτά έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και άρα πρόκειται περί παραβίασης της συνθήκης και του δικαίου. Τώρα, τι θα γίνει όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφοριών, την αντιτρομοκρατική προσπάθεια, γιατί είπαμε ότι αν έχουμε hard Brexit, τότε τι θα γίνει με την ε, συνεργασία στο επίπεδο αυτό της αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Φαίνεται πλήγμα μεγάλο το να μην μπορούμε να έχουμε πλήρη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες της ε, Βρετανίας. Τι γίνεται, ε, όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα ε, προεκλογικά ή έχουν κάποια βάση. Ελπίζω να δούμε, ξεκαθαρίσουμε τι θα ισχύσει από πρώτα ουσίας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Γκί. Θα ξεκινήσω από τις διαφορετικές ερωτήσεις όχι θα προσπαθήσω να τις βάλω σε ομάδες. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν ρωτήσει για το ίδιο θέμα. Κάποιοι μίλησαν για την Ιρλανδία και την Βόρεια Ιρλανδία. Ε, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, για παράδειγμα, της Μεγάλης Παρασκευής, Good Friday Agreement. Και από τις δύο πλευρές συμφωνούμε να εφαρμόσουμε πλήρως τη συγκεκριμένη συμφωνία στο μέλλον. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν την συνέχιση της συμφωνίας αυτής των αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Βόρειας Ιρλανδίας που έχουν Ιρλανδικό διαβατήριο. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε λοιπόν όλα τα δικαιώματα που τους ε, παραχωρεί το ε, διαβατήριο αυτό. Ε, Μακίνες είπε ότι μία λύση είναι να μείνει στην ε, Τελωνιακή Ένωση και την κοινή αγορά. Συμφωνώ προσωπικά, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζήτημα που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά μας στις αρχές Οκτωβρίου πρόθεσή μου είναι λοιπόν να υπάρξουν τουλάχιστον κάποιες παράγραφοι στο κείμενο που να αφορούν στο ζήτημα αυτό που έθιξαν ο κ. Άνδρος και κυρία Μαγκίνες. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στις οικονομικές αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της James και του κυρίου Μπάτν. Εγώ δεν έκανα λόγο για ηθικές υποχρεώσεις χρησιμοποίησα τα λόγια του κυρίου Ντέιβις όταν ανέφερα τον όρο ηθικές υποχρεώσεις. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει νομική βάση φυσικά και η νομική βάση αυτή είναι σαφής στα έγγραφα, στα έγγραφα που έχει α, ήδη συντάξει, έχει προωθήσει ο κύριος Μπαρνιέ. Είναι δημόσια τα έγγραφα αυτά, ο καθένας μπορεί να τα συμβουλευτεί και υπάρχουν αρκετά άρθρα τα οποία περιγράφουν πού ακριβώς βασίζονται αυτές, οι οικονομικές αποπληρωμές. Συγχωρέστε με, αλλά δεν θα υπησέλθω σε μια συζήτηση που αφορά στο πόσα δισεκατομμύρια είναι οι οικονομικές αποζημιώσεις. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι διαπραγματευτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ποτέ δεν έθεσαν το ζήτημα σε συζήτηση. δεν ξεκίνησαν μια συζήτηση σχετικά με το αν υφίστανται ή όχι. Σεβόμαστε την διάσταση. Σεβόμαστε τη συζήτηση αυτή, με συγχωρείτε, και βεβαίως σε ό,τι αφορά τους όρους των μειώσεων για την Μεγάλη Βρετανία. Ένα άλλο ζήτημα αφορά στα δικαιώματα των πολιτών. Κάποιοι συνάδελφοι τα έθιξαν. Ε, κυρία Μπρεσό, έχω συζητήσει μαζί της. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα αυτή θα πρέπει να μεταφραστεί σε μια διεθνή συμφωνία. θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα, αν το δικαστήριο δεν αρκεί, δεν θα είναι ένα μονομερές σύστημα όμως. Γι' αυτό και κάνουμε λόγο για μια διεθνή συμφωνία. Και όχι, και όχι μόνο μια μονομερής νομοθεσία από πλευράς Βρετανίας που μπορεί να την αλλάξει το Βρετανικό Κοινοβούλιο ανα πάσα στιγμή. Φτάνω τώρα στο επόμενο σημείο μου. Νομίζω ότι ήταν η Μπάρμπαρα Σπινέλη που έθιξε το ζήτημα αυτό. Θυμάστε πολύ καλά την ορολογία που χρησιμοποίησαμε εμείς στο δικό μας ψήφισμα. Διάβασε το ξανά γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι σημαντική Είναι ανάγκη να το επαναλάβουμε. Γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία, θα είναι πολύ κοντά το κείμενο σε αυτό που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Μπάρμπαρα και άλλοι έκαναν λόγο για αυτήν την λεγόμενη μεταβατική συμφωνία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες φωνές, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και εδώ, που κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας μεταβατικής συμφωνίας. Δεν είναι μόνο η εργατική, αλλά και μεμονωμένα μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και του κυβερνώντος κόμματος για μας δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει γιατί και εμείς ως κοινοβούλιο από την πρώτη κιόλας μέρα κάναμε λόγο για μια μεταβατική περίοδο που θα είναι αναγκαία. Γιατί, γιατί όλοι μας έχουμε μια ελάχιστη εμπειρία. Ξέρουμε ότι εδώ και ε, μάλλον στον επόμενο χρόνο, ένας χρόνος και ένας μήνας που μας περισσεύει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τη μελλοντική μας συνεργασία, σχέση και τα βήματα για να φτάσουμε σε αυτή την μελλοντική σχέση. Και εμείς αυτό το είπαμε από την πρώτη κιόλας μέρα στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό έχουμε ήδη ε, θίξει την ανάγκη μιας μεταβατικής περίοδου, αλλά και να θέσουμε τα χρονικά πλαίσια της μετα... μεταβατικής αυτής περίοδου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τώρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θυμάμαι ένα χρόνο πριν, στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλοί ισχυρίζονταν ότι μέσα σε δύο χρόνια θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τα πάντα. Ε, θεωρώ ότι εμείς ήμασταν πολύ πιο ρεαλιστές ως κοινοβούλιο να συζητάμε από την πρώτη κιόλας μέρα για την ανάγκη δημιουργίας μιας μεταβατικής συμφωνίας. Η οπτική μας γωνία, κυρία Σπανέλη, όταν, Σπινέλη, όταν κάνουμε λόγο για μεταβατική περίοδο, είναι η συνέχιση αυτού που έχουμε σήμερα και μια σταδιακή αποχώρηση. Είναι αδύνατον να έχουμε κάτι εντελώς καινούριο και να το ονομάσουμε μεταβατικό. Το μεταβατικό είναι αυτό που έχουμε που σιγά σιγά θα αποδυναμώνεται σταδιακά. Ας είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το τι είναι δυνατόν. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια μεταβατική περίοδο και η μεταβατική αυτή συμφωνία θα πρέπει να είναι λίγο έως πολύ αυτό που ισχύει σήμερα τα σημερινά και, και εκτιμένα τα οποία σιγά σιγά σιγά σταδιακά θα αποδυναμώνονται. Και αυτό με φέρνει στο επόμενο ζήτημα που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Θεωρώ αυτό που πρέπει να κάνουμε να επιταχύνουμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών να συμφωνήσουμε σε κάτι που ξέρουμε ότι στο τέλος θα είναι κομμάτι της γενικής συμφωνίας. Θεωρώ ότι πρέπει να επιταχύνουμε στο σημείο αυτό. Και οι δύο πλευρές από κοινού να δημοσιεύσουμε αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά τα οποία αποφασίζουμε Να ξέρουμε όμως ότι επισήμω αυτό θα είναι κομμάτι της τελικής συμφωνίας αποχώρησης. Κύριε Άντερσον, τώρα ε, ε, σε ό,τι αφορά το πόσο ικανή είναι η κυβέρνηση των Τόρι ή όχι, δικό σα είναι αυτό που είπατε. Έτσι, εσεί αναλαμβάνετε την ευθύνη, γιατί μπορώ εύκολα να φανταστώ να αναφερθεί κάτι στον τύπο αύριο το Βρετανικό. Αλλά ε, όταν έδωσα την απάντησή μου στην ε, Μπάρμπαρα Σπινέλη, ε, είπα ότι σε αυτήν την συμφωνία σε ό,τι αφορά την ε, μεταβατική, ή μάλλον είναι σαφές στη συμφωνία πλέον ότι θα χρειαστεί μια μεταβατική περίοδο, περίοδος και Νομίζω πως ε, ε, δεν υπάρχει αμφισημία και από την πλευρά του. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα σε σχέση με τα ζητήματα εμπορίου. Εδώ το ζήτημα είναι ότι μόλις λάβει χώρα επίσημη αποχώρηση, δεν αποτελεί πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο επίσημο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και κατά συνέπεια έχει τη δυνατότητα πλέον να προβεί σε δικές του ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες. Και εμείς είπαμε ότι στο μεταξύ και είμαστε το μοναδικό θεσμικό όργανο που το έκανε. Είπαμε λοιπόν στο μεταξύ σε δικό μας ψήφισμα ποια είναι η δική μας άποψη ως προς τις δυνητικές συνέπειες σε σχέση με ε, συμφωνίες οι οποίες τη χάνουν ε, πριν ακριβώς από την επίσημη αποχώρηση. Γιατί βέβαια εδώ βασιζόμαστε στην αρχή ότι δεν μπορεί κανείς ε, να έχει και τα δύο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις ξεχωριστές διμερείς με μια χώρα και από την άλλη πλευρά να συμμετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις τις οποίες θα κάνει δηλαδή εξ ονόματος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση με αυτή τη χώρα. Ε, δεν αναφέρεται ωστόσο κάτι τέτοιο στις κατευθυντήρες γραμμές του Συμβουλίου ή κάπου αλλού. εμείς ως Κοινοβούλιο το αναφέραμε στο ψήφισμά μας, Δηλαδή, ποιε θεωρούμε ότι θα ήταν οι συνέπειες ε, στο πλαίσιο τέτοιων ε, συμφωνιών. Τώρα, κύριε Καστάτο, νομίζω πως ε, ε το Κοινοβούλιο προς το μέλλον έχει πει ξεκάθαρα τι επιθυμεί. Θέλουμε μια συμφωνία σύνδεση. Και γιατί? Ε, γιατί πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο απαντάται στη συνθήκη, ένα νέο εργαλείο το οποίο έχει προβλεφθεί ω νέο εργαλείο στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και από εκεί και μετά, επειδή αυτή η συμφωνία σύνδεση ε, παρέχει μεγάλα περιθώρια ευελιξία. Μία δηλαδή συμφωνία σύνδεση ε, μπορεί να είναι περιορισμένη, αλλά μπορεί να είναι και μια ευρεία συμφωνία. Ε, μπορεί να αφορά μόνο εμπορικά ζητήματα, αλλά μπορεί να αφορά σύνδεση σε ό,τι αφορά τομείς όπως αυτός της έρευνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας αλλά και άμυνας εξωτερική δηλαδή ασφαλεία. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τάχθηκε υπέρ της ε, συμφωνίας ε, σύνδεσης ως η ε, καλύτερη μελλοντική συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά προφανώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη φάση. Προσπαθούμε σε αυτή τη φάση ακόμα να ολοκληρώσουμε ε, τα τη αποχώρηση. Τώρα, ε, σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Κόρμπετ ε, σε ό,τι αφορά ε, την, το ποιο κατηγορεί ποιον και πράγματι εγώ εκπλήσωμαι με τα άρθρα που διαβάζω μερικέ φορέ ω προ τι ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη η οποία αποφάσισε να διώξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το αντίθετο. Ακριβώ το ανάποδο έλαβε χώρα. Οπότε ε, αυτή η απόφαση ήταν ανεξάρτητη και αυτόνομη ε, για αποχώρηση από την πλευρά ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και βέβαια εξακολουθεί να με λυπεί η απόφαση αυτή. Καλώς. Νομίζω πως εξαντλήσει και η συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα εκεί όπου να επανέλθει στη δική μας συνεδρίαση προφανώς είσαι θέμα προσκεκλημένος. Ναι, νομίζω πως ε, θα ήταν καλό να επανέλθω όταν θα έχουμε την πρόσταση ψηφίσματος από την πλευρά της ΑΦΚΟ. Άρα, συνάδελφοι, έχουμε ακόμα τα διάφορα στην ημερήσια διάταξή μας. Δεν υπάρχουν διάφορα από την πλευρά κανένας συναδέλφου και η συνεδρίαση για την επόμενη συνεδρίαση. Έχουμε 11 Σεπτεμβρίου μια έκτακτη συνεδρίαση και από εκεί και μετά 28 ε, Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση. Οι συντονιστές σας παρακαλώ να παραμείνετε μέσα στην αίθουσα για να συνεχίσουμε κατευθείαν με τη δική μας συνεδρίαση.